ότι πολλές από τις αποφάσεις δεν ήταν τόσο καλές όσο θα θέλαμε. Να σας θυμίσω στον Ντέρμπαν, όλα τα μέρη δήλωσαν ότι δεν ήταν έτοιμα να κάνουν μια σημαντική συμφωνία πριν το 2015. Και η διαδικασία αυτή δεν εκπλήσει κανέναν. Ξαφνικά επιταχυνόμενοι πρέπει να έχουμε ρεαλιστικές, είχαμε ρεαλιστικές προσδοκίες για, ε, για την έκβαση της ε, Βαρσοβίας. Πιστεύω ότι καταφέραμε να χειριστούμε τη χρηματική πλευρά με αξιοπρεπή τρόπο. Πολλά κράτη-μέλη ουσιαστικά πρότειναν χρηματοδότηση που καταδεικνύει ότι βρισκόμαστε σε ε, φάση βελτίωσης όσον αφορά τη χρηματοδότηση στην Ευρώπη. Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, πιστεύω ότι η έκβαση ήταν αρκετά ικανοποιητική. Σημειώσαμε σημαντική πρόοδο για τις απώλειες και τις ζημίες, αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για τις πιο ευάλωτες χώρες εδώ και 20 χρόνια. Βλέποντας τι έχει γραφτεί και στο δικό τους τύπο, όταν γύρισαν στις χώρες τους θεώρησαν ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Αυτή η αντιμετώπιση σημερινή των απολειών και των ζημιών χωρίς ε, να δημιουργείται μια σειρά νέων θεσμικών θεσμών. Το βασικό ζήτημα το Σάββατο φυσικά ήταν το ADP. Το πρόγραμμα δηλαδή από τώρα μέχρι τη διάσκεψη του Περισσίων. Αυτό που ζητήσαμε είναι ότι θέλαμε ένα χρονοδιάγραμμα και το πήραμε. Είπαμε ότι όλοι θέλουν, ε, έχουν κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε μέχρι το 2014. Καταλήξαμε στο πρώτο τρίμηνο του 2015 και για, φυσικά για όποιους ήταν έτοιμοι δεν μπορούμε να υπαγορεύσουμε, να επιβάλλουμε σε όλους να κάνουν τη δουλειά στα εθνικά του κοινοβούλια αν δεν το επιθυμούν. Αλλά αποφασίστηκε ότι μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2015 θα πρέπει να έχουμε τα διάφορα σχέδια ε, από τις διάφορες χώρες ώστε έγκαιρα πριν το Παρίσι να μπορούμε να δούμε κατά πόσο η συνδυασμένη προσπάθεια θα βοηθήσει όλο τον κόσμο να παραμείνει κάτω από τους δύο βαθμούς. Είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη να υπάρξουν αυτές οι δυνητικές υποσχέσεις αρκετό καιρό πριν το Παρίσι. Για ποιο λόγο? Διότι αυτό κάνει τη διαφορά μεταξύ ενός καθεστώτος από κάτω προς τα πάνω όπου απλά έρχεται ο καθένας και λέει τι θέλει και το υβριδικό ε, σχέδιο προσπαθούμε να φτιάξουμε από πάνω προς τα κάτω όπου η προσέγγιση από bottom-up δεν θα επιτύχει αρκετά αποτελέσματα. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, ένα ευρυδικό πρόγραμμα και πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα σχέδια της κάθε χώρας ώστε να μπορέσουμε στη διεθνή κοινότητα να συζητήσουμε και να δούμε εάν δεν επιτυχάνονται τα αποτελέσματα που θέλουμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αυτό πιστεύω ήταν πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι οι Γάλλοι συνάδελφοι πρέπει να είναι αρκετά ικανοποιημένοι γιατί τώρα έχουν ε, υλικό στο οποίο μπορούν να εργαστούν και όσοι ήταν εκεί μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι η πολύ σημαντική συζήτηση, η πιο σημαντική συζήτηση ήταν σαν να βρισκόμαστε ξανά πίσω στον Τέρμπαν. Υπήρξαν κάποιες χώρες που προσπάθησαν να οπισθοχωρήσουν. Δεν το επέτυχαν. Και τι κάνουμε εδώ. Όλοι θεωρούμε ότι πρέπει να είναι εξίσου νομικά δεσμευμένοι όπως έγινε στο Τέρμπαν. Μην ξεχνάμε ότι αυτά που ε, βιώσαμε στη Βαρσοβία δείχνουν πόσο δύσκολο ήταν ο δρόμος μέχρι το Παρίσι. Η θετική πλευρά είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε συμμετείχαν περισσότερο στι συνομιλίε και δεσμεύτηκαν περισσότερο από ό,τι έχουμε δει εδώ και καιρό και ανακοίνωσαν δημόσια ότι είναι έτοιμε στο πρώτο τρίμηνο του 2015 να μα ανακοινώσουν τι προθέσει του. Κάποια καλά πράγματα λοιπόν, καλά αποτελέσματα προέκυψαν και θα θυμάστε ορισμένοι από εσά ότι είπαμε πως είναι σημαντικό του χρόνου να έχουμε αποφασίσει όσοι βρίσκονται στη δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του Κιώτο να έχουν αποφασίσει ήδη πώς θα αναθεωρήσουν τι πρόκειται να κάνουν από τώρα μέχρι το 2020. Για προφανείς λόγους θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ σημαντικό η άσκηση αυτή για το πώς θα ε, καταλήξουμε στο τι θα κάνουμε μέχρι το 2020 θα πρέπει να αφορά όλες τις χώρες. Και αυτό αντικατοπτρίζεται πολύ σαφώς και στην απόφαση της Βαρσοβίας ότι τον Ιούνιο του χρόνου θα γίνει μια υπουργική διάσκεψη όπου όλα τα μέρη είτε ανήκουν στην ε, δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του Κιώτο είτε όχι θα συμμετάσχουν σε αυτή την υπουργική διάσκεψη όπου θα συζητήσουμε τι θα κάνουμε σε αυτή τη φάση μέχρι το 2020. Τελευταίο σημείο. Στο, αναφέρθηκαν δεσμεύσεις για, και δράσεις με οικονομική δράση για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτή είναι η γλώσσα του Κιώτο. Εμείς θα θέλαμε κάποιες δεσμεύσεις όπως τις ζητάμε για όλους αλλά υπήρξε κάποια αντιπαράθεση σε αυτό, αλλά πετύχαμε τη λέξη contribution, συμβολές, αλλά με πολύ σαφή αναφορά μετά από αυτή τη λέξη ότι αυτό δεν προδικάζει τη νομική μορφή των ε, δεσμεύσεων αυτών. Και το σημαντικό είναι ότι τουλάχιστον τώρα ξεφορτωθήκαμε αυτά στις διαφορετικές δεσμεύσει για τις ε, αναπτυγμένες και άλλες δεσμεύσει για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Όλοι πρέπει πλέον να συμμορφώνονται με τα ίδια. Αλλά φυσικά ε, πρόκειται η συζήτηση να είναι μακροχρόνια όσον αφορά την νομική μορφή αυτών των συμβολών. Συνολικά κύριε Πρόεδρε ήθελα να πω ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Η επερχόμενη γαλλική προεδρία τώρα έχει ένα χρονοδιάγραμμα μπροστά της και η στρατηγική μας ε, θα βασιστεί σε μια σειρά βημάτων και πιστεύω ότι αυτό ήταν η καλή έκβαση της διάσκεψης τελικά. Ευχαριστώ Κόνι Χέντεγκαρτ και, και για τη συνόψη για τη Βαρσοβία. Προσωπικά και μίλησα και με κάποιους που ήταν ε, παρόντες προέκυψαν περισσότερα από όσα περιμέναμε. Υπήρχαν κάποιες ε, παραφωνίες ότι θα πρέπει να είναι πιο επιτυχημένη η οργάνωση. Χρειάστηκε μια ολόκληρη μέρα για να το οργανώσουμε όλα αυτά. Δεν ήταν τόσο αποτελεσματική οργάνωση, πρέπει να το πω. Αλλά εν ήταν κάτι που μπορεί να μας ικανοποιήσει, ένα μικρό βήμα μπροστά, σαν τυχελό να πηγαίνει η περιβαλλοντική πολιτική, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα βήμα μπροστά. Δεν έγινε τουλάχιστον καμιά καταστροφή. Γιατί έχουν γίνει και καταστροφές για τις εκπομπές ε, από την αυτιλία. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Υπάρχει ε, ένας τομέας όπου έχουμε τεράστια κρίση, τα ναυπηγεία. Θα μπορούσε να είναι αυτό ένα συγκυριακό πρόγραμμα για τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία. Αν μειώσουμε κατά 70% με τεχνικά μέτρα, ε, κατά 75% όπως έλεγα λοιπόν, ε, τις εκπομπές. Έχουμε κάτι πολύ θετικό για ε, τα λιμάνια μας, διότι εκεί επειδή ε, κοντά στα λιμάνια φυσικά χρησιμοποιείται τόσο πολύ καύσιμο, υπάρχουν πολλά προβλήματα με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Είναι λοιπόν θέμα όχι γενικά περιβάλλοντος, αλλά και πιο συγκεκριμένα ποιότητας του αέρα. Είχαμε με την έκθεση χάσει όπου αναφερθήκαμε και στην ποιότητα των ε, καυσίμων. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε τα δύο νομοθετήματα να μην αντιπαρατίθενται. Γιατί και αυτό και έχει υπάρξει για κάποια μέτρα ε, για τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν όμως οι τεχνολογίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα ε, ξεπεράσουμε. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε και η Κομισιόν και όλοι οι άλλοι, θα πρέπει ώστε να τον πιο έγκαιρα, να έχουμε αυτά τα νέα πλοία ε, που είναι πολύ πιο περιβαλλοντικά. Υπάρχει ούτως ή άλλως τεράστιο υπερβολικό δυναμικό. Αν πάει κανείς στα λιμάνια θα δείτε ε, πόσα ε, πλοία εμπορευματοκιβωτίων είναι αραγμένα. Θα πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή μέσω, μέσω μείωσης της, ε, μείωσης ε, της ε, του δυναμικού αυξάνονται βεβαίως οι ναύλοι. Άρα βελτιώνεται η κατάσταση. Και έτσι τελικά βελτιώνεται και η οικονομία και το κλίμα γενικά και η ποιότητα του αέρα. Αν δεν κάνουμε τίποτα, αν συνεχίσουμε όπως έχουν τα πράγματα, business as usual, θα ανεβούν από το 2010 έως το 2020 κατά 50, 51% εκπομπές από την αυτιλία. Άρα πρέπει να το κάνουμε, έχει έννοια να το κάνουμε. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε αυτή τη συζήτηση και θα ε, ε, επιτύχουμε πιστεύω σημαντικά. Λοιπόν, οι συντονιστές πρώτα απ' όλα, Ζέμπερ, μετά Μακάβαν και μετά ο Chris Davis. και ο κύριος Κυλακάκης θα μιλήσει αντί του Chris Davis, ο οποίος είναι εισηγητής ε, για το επόμενο θέμα που ε, σχετίζεται. Αλλά πρώτος ο, Ρίχαρτ Ευχαριστώ Ματίας. Να ξεκινήσω με την αυτιλία. Όπως είδαμε και στις αερομεταφορές, είναι πολύ δύσκολη τομή αυτή όπου υπάρχουν, ε, υπάρχει αυτή η παγκόσμια διάσταση θα πρέπει να ξεκινήσει με τη συλλογή στοιχείων η Κομισιόν. Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Αλλά πιστεύω ότι επίσης θα πρέπει να έχουμε μια νέα προσέγγιση, όχι μόνο συντρογή στοιχείων, μετά μέτρα ε, με βάση την αγορά. Αυτό κάνουμε σε άλλους τομείς. Νομίζω ότι στον τομέα αυτό, όπως και στον ε, τομέα τον αεροπορικό, είναι πολύ δύσκολο γιατί υπάρχει διεθνής ανταγωνισμός και σχετίζεται με τις εκπομπές άνθρακα carbon linkage με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ωραία, βεβαίω σωστά να συλλέξουμε στοιχεία και μετά να δούμε τι θα κάνουμε περαιτέρω, όπως είπε και ο Ματίας ο Πρόεδρος, να δούμε τι θα κάνουμε, ούτω ώστε αυτές οι τεχνολογικές αλλαγές να φτάνουν πολύ γρήγορα στην αγορά. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Διότι υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες επιτρέπουν τεράστιες εξοικονομήσεις διοξιδίου του άνθρακα και άλλων ρηπαντών και έτσι θα επιτύχουμε τα πλοία μας. Ε, μάλλον το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα επιτύχουμε να ε, επανεξοπλίσουμε τα πλοία μας. Αλλά τα μέτρα αυτά έχουν το αποτέλεσμα ότι μειώνουν το δεξίδο του άνθρακα από τη μία, άρα καλύτερος αέρας, ε, λιγότερη κατανάλωση, πολύ θετικά αποτελέσματα. Και από την άλλη πλευρά δεν μας δημιουργούν πρόβλημα με τους διεθνείς εταίρους μας και επιπλέον τρίτον έχουμε τη δυνατότητα να πουλήσουμε αυτά τα νέα σύγχρονα πλοία στη διεθνή αγορά. Παίρνουμε λοιπόν μέτρα τα οποία έχουν πολλαπλή θετική δράση, βοηθάνε συνολικά τον τομέα μας. Έχουν έννοια και δεν μας δημιουργούν προβλήματα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρακαλώ λοιπόν την Κομισιόν να δει μια πολύ θετική αντιμετώπιση για πρώτη φορά σε αυτό το τομέα. Να μην συνεχίσουμε με την παλιά προσέγγιση, στόχοι, μηχανισμοί, μέτρα, γιατί μας δημιουργούν δυσχέρειες, όπως είδαμε και στις αερομεταφορές. Όλη η συζήτηση για την κρυφοκρατία και τα α και τα β τη γνωρίζουμε. Πρέπει να είμαστε κάπως καινοτόμοι, να επιδιώξουμε, να δούμε με άλλα γυαλιά. Για τις διαπραγματεύσεις στη Βαλσοβία δεν ήμουν παρόν. Είναι μια επιτυχία που επετεύχθη με μικρά βήματα. Το βασικό είναι να συνεχίσουμε. Να μην ε, σταματήσουμε την πορεία, να μην βαλτώσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία μακροπρόθεσμα έναντι της κοινή γνώμης, διότι ξέρετε λόγω της οικονομικής κατάστασης ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για την περιβαλλοντική πολιτική, αλλά μακροπρόθεσμα οπωσδήποτε θα γίνει θέμα. Πρέπει λοιπόν, βεβαίως ξέρουμε τις δυσχέρειες που έχουν ε, οι αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα με την ποιότητα του αέρα, αλλά θα γίνει για όλους μας θέμα, γιατί οι εξελίξεις αυτές πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος ημών. Δεν είναι το θέμα ε, βέβαια να εμφανιστούμε στα μέσα ως ε, αυτοί που κέρδισαν τα πολλά. Ξέρετε ότι τα μέσα πάντα θέλουν να λένε Κάποιοι πέτυχαν, κάποια απέτυχαν. Το θέμα είναι να επιτύχουμε τους στόχους όμως. Πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να σημειωθεί περαιτέρω προόδος, να δείξουμε αντοχή, μακροπρόθεσμα, να επιτύχουμε να μην ξεπεράσουμε τους δύο βαθμούς, αλλά πιστεύω ότι αυτή η διάσκεψη ήταν λοιπόν ένα βήμα προς την καλή κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν να αρκεστούμε στον δεν υπήρχαν μεγάλες πρόοδοι, αλλά νομίζω ότι η κοινή γνώμη θα συνεχίσει να παίζει ένα ε, θετικό ρόλο και ε, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να την έχουμε με το πλευρό μας. Παρακαλώ λοιπόν την Κόνη να συνεχίσει να εκπροσωπεί τόσο πολύ ε, σωστά και με αρκετή φιλοδοξία την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Βεβαίως και αυτό πρέπει να υποθεί, ο πρόεδρος. Ωραία. Μακάβαν. Ε, λοιπόν, κλείνω τον κατάλογο των ομιλητών. Λίντα Μακάβαν, λοιπόν, ε, μετά ο συνάδελφος Σκυλακάκης, Ρόσμπαχ, Σιμάνσκι, Φλόρεντς, Γιόρξεν και Γκεμπράντι. Ξέχασα κανέναν. Ωραία. Κλείνω το κατάλογο λοιπόν. Μακάβεν. Ευχαριστώ Κόνη για όλες τις πληροφορίες. Συνεχίζεται το έργο, αυτό έχει σημασία. Συνεχίζεται όλη αυτή η διαδικασία. Μα αφείτε. Οπότε το χρονικό πλαίσιο των, ε, της επόμενης διάσκεψης στο Παρίσι δεν θα είναι εύκολη συγκυρία γιατί θα είμαστε και ένα έτος πριν από τις ε, αμερικανικές εκλογές και δύσκολα θα καταφέρουμε να δεχθεί και ο πρόεδρος τον ΗΠΑ ε, κάτι το οποίο με πολύ μεγάλη δυσκολία θα περάσει από το Κογκρέσο. Το ίδιο Μπορεί να συμβαίνει και στην Επιτροπή, αλλά δηλαδή να υιοθετείται μια νομοθετική πρόταση, όμως δεν χρειάζεται να το φτάσουν μέχρι τέλους στη δική μας περίπτωση. Και στο Κοινοβούλιο είναι πιο δύσκολα τα πράγματα σε αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα. Το ξέρει και ο Ρίτσαρντ, ε, όλο ένα και μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε και στην Ολομέλεια βλέπουμε αυτές τις δυσκολίες. και στο Συμβούλιο αλλά και στη χώρα μου υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για ε, το περιβάλλον και τα ζητήματα οικολογίας και πιο συγκεκριμένα για το κόστος ε, και την δομή αυτής της πολιτικής. Κάποιες τέτοιες αποφάσεις είχαν ληφθεί ε, όταν υπήρχε υπόθεση της συνεχούς ανάπτυξης. Τώρα έχουμε νέους στόχους που δεν θα είναι εύκολη συζήτηση ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο μάλλον ε, ευρύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, μήπως θα πρέπει να αλλάξει όμως λίγο την ορολογία της, αν θέλετε, ή και γενικότερα τα επιχειρήματά της. Υπάρχουν πολλές, πολλές υπερβολές στο αφορά το κόστος ε, της πράσινης ενέργειας, όμως ε, ισχύει ότι κάποιες πτυχές είναι πράγματι ότι ο καταναλωτής είναι αυτός που ε, επομίζεται το κόστος ε, αυτής της ενέργειας. Πώς ε, συμπεριλαμβάνεται τη διάσταση της προσβασιμότητας των τιμών. Δηλαδή, σε πολλές χώρες δεν έχουμε επενδύσει σε έργα μόνος για παράδειγμα, γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι οικονομικές περικοπές και περιορισμοί. Τι θα γίνει λοιπόν, ιδάλλως δεν υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθείτε ως ένας οργανισμός που αυξάνει το κόστος, δεν βρίσκει ρεαλιστικούς τρόπους να μειωθεί το κόστος αυτό και μετά τελικά θα φτάσουμε το 2015 και δεν θα έχουμε ούτε καν εμείς κάποιους ρεαλιστικούς στόχους ε, για το 2030. Αυτό με βάση τη δική μου εμπειρία, τη δική μου χώρα, αλλά νομίζω δεν αλλάζει η κατάσταση αλλού. Well, uh, uh, Ως εισηγητής, θα επικεντρωθώ κυρίως ε, στο ζήτημα του MRV, ε, τη παρακολούθηση υποβολή εκθέσεων και επαλήθευσης, που είναι σημαντικό θέμα κατά τη γνώμη μου. Αρχικά, θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό ε, να μετρούμε επακριβώς και εκτεταμένα όλα, όλους τους σημαντικούς ε, όλα τα αέρα του θερμοκηπίου ε, τα οποία εκπέμπουν τα πλοία. Αυτό προσπάθησα να κάνω και στη δική μου έκθεση. Με την επέκταση του πεδίου εφαρμογή. Όμως ε, είναι σημαντικό αυτό να γίνεται και με έναν κάτω το δυνατόν αποδοτικό και συναφή τρόπο. Ένας φίλος μου που τον χώρο της δημοσιογραφίας μου είπε κάποια στιγμή μην αφήνεις την πραγματικότητα να σου καταστρέψει, να σου αχρηστεύσει ένα καλό επιχείρημα. Δυστυχώς θα πρέπει αυτό όμως να κάνω σε ό,τι αφορά τις εκπομπές των πλοίων για να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνουμε. Αν διαβάσετε την αξιολόγηση αντικτύπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος ε, σε ό,τι φορά τα πλοία και την ατμόσφαιρα, είδαμε ότι μέχρι το 2020 τα πλοία έχουν αρνητική επίπτωση σε διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά ε, τα αέρια του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό είναι ένα μικρό τμήμα της πραγματικότητας που πρέπει όμως να το λάβουμε υπόψη. Αυτό βεβαίως και θα αλλάξει για δύο κυρίως λόγους γιατί πρώτον θα αυξηθεί η εμπορική δραστηριότητα στα επόμενα 30 χρόνια σε πολύ μεγάλο βαθμό και το θαλάσσιο εμπόριο που είναι ο πιο αποδοτικός ε, τρόπος μεταφορών επίσης θα αυξηθεί πολύ. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι θα υπάρξει αύξηση. Και ε, η ρήπη που σε τοπικό επίπεδο ε, λειτουργούν αρνητικά, όμως σε διεθνές επίπεδο όχι, θα αυξηθούν επίσης. Μέχρι λοιπόν το 2020 έχουμε ε, ακόμα έναν παγκόσμιο αντίκτυπο ε, ψήξης, η μείωση της θερμοκρασίας. Μετά από εκεί όμως θα περάσουμε σε αρνητικό αντίκτυπο που θα αυξηθεί με τον καιρό. Επίσης υπάρχουν δυνατότητες για την εξοικονόμηση και την αύξηση της ενεργικής απόδοσης, όμως ο Διεθνής Αυτιλιακός Οργανισμός, ο IMO, από όπου αντλεί και τα δεδομένα της Κομισιόν, δεν λέει μέχρι 75%. Μιλάει πιο συγκεκριμένα, λέει 25 έως 75%. Επομένως, αυτή είναι η πραγματικότητα. 25 με 75%, όχι έως 75%. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικά ωφέλη, τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε, αλλά πρέπει να τα μετρήσουμε με ρεαλιστικό και αποδοτικό τρόπο. Να σημειώσουμε επίσης ότι τα δύο τρίτα του κόστους ενός ε, ε, πλοίου είναι τα καύσιμα. Πολύ σημαντικά κίνητρα υπάρχουν λοιπόν για να είναι ένα πλοίο ενεργειακά αποδοτικό. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν μπορεί να συμβεί γιατί σε όλες τις επιχειρήσεις η αποδοτικότητα ως προς την αγορά είναι αυτό που τις ενδιαφέρει. Εμείς πρέπει να διορθώσουμε ανεπάρκειες της αγοράς και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να μετρούμε τις, ε, τα αέρια του θερμοκηπίου και να τα τιμολογήσουμε στο μέλλον, κατά τη γνώμη μου. Με ένα τέλος, κατά τη γνώμη μου. Γιατί αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα ETS ε, σε παγκόσμιο επίπεδο δεν πρόκειται αυτό να λειτουργήσει. Αυτό είναι άλλη συζήτηση όμως. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα, θεωρώ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο δυνατόν πιο κοντά στο αμερικανικό σχέδιο το οποίο έχει προταθεί στον IMO, το οποίο είναι ένα καλό σχέδιο και έτσι να έχουμε ένα πολύ εύρωστο επιχείρημα και να έχει λόγο και ο IMO να προχωρήσει με το σύστημα παρακολούθησης ε, και υποβολή εκθέσεων και το καθεξής. Γιατί αν είναι μόνο ευρωπαϊκό αυτό το σύστημα δεν ε, ε, θα λύσουμε το πρόβλημα. Η ναυτιλία είναι η πιο παγκόσμια ο πιο παγκόσμιος καθολικός κλάδος της επιχείρησης, ε, του επιχειρηματικού κόσμου μπορείτε να φανταστείτε. Αλλάζουν δρομολόγια, αλλάζουν τόπο δραστηριοποίησης. υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορεί να επιλέξουν έναν ε, κόμβο ε, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ιδίως στη Μεσόγειο συμβαίνει αυτό. Πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε το πεδίο εφαρμογή και για τα μικρά πλοία και να πέσουμε στα 400 όπως προτείνει η Αμερικανική πλευρά αυτή τη στιγμή στον IMO και να κρατήσουμε αυτή την πρόταση ως δυνατόν απλούστερη για να διευκολύνουμε και το Συμβούλιο και τον Διεθνή Αυτελειακό Οργανισμό για να ε, προχωρήσει αυτός ο φάκελος το συντομότερο δυνατόν. Θεωρώ ότι έχουμε χρόνο να ολοκληρώσουμε αυτό το φάκελο και πραγματικά θα ήθελα να επιτευχθεί αυτό και έτσι να συμβάλλουμε στη θέσπιση ενός παγκοσμίου MRV. Με τα διαχειριστικά σχέδια ενεργειακής απόδοσης των πλοίων ε, είναι μια πολύ σημαντική κίνηση ε, που υιοθέτησε ο IMO. Η ενεργειακή απόδοση και στο σχεδιασμό είναι θετικό βήμα. Εάν προσθέσουμε και ένα διεθνές MRV, φτάνουμε πολύ κοντά στο επόμενο βήμα αυτής της ε, συνολικής διαδικασίας. Αυτά ήθελα να πω. Μια σύντομη παρατήρηση ακόμα για τις ε, διαπραγματεύσεις για το κλίμα. πρέπει να λάβουμε υπόψη και την οικονομική κατάπτωση, που είναι μια πραγματικότητα. Για πολλά χρόνια πλέον έχουμε χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από, από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και σε σχέση με την ανάπτυξη που εμείς είχαμε προβλέψει στην έναρξη της πολιτικής. Και όλα αυτά αλλάζουν τους υπολογισμούς μας πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό στα επιχειρήματά μας. Δεν είμαστε πλέον η πλούσια και ισχυρή ε, ήπειρος που μπορεί γενναιόδωρα ε, και με μεγαλοψυχία να βοηθήσει τους πάντες. Έχουμε πολύ ψηλή ανεργία, βρισκόμαστε σε βαθιά οικονομική κρίση και δεν είναι κρίση του κόσμου, αλλά της δύση και ιδίως της Ευρώπης. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό. Μόνο ένα παράδειγμα θα σας αναφέρω. Στη χώρα μου, στην Ελλάδα, μείον 25% του ΑΕΠ. Τώρα, οι εκπομπές κατά κεφαλήν είναι κατά πιθανότητα στο ίδιο επίπεδο, ίσως και λιγότερες, από τις εκπομπές κατά κεφαλήν στην Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει καμία όμως απολύτως υποχρέωση στην πραγματικότητα λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα. Ιδίω με του γειτονέ μα και πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι αναφερόμεθα σε πολλά θέματα, αλλά παρακαλώ τους συναδέλφου να τηρούν ε, κάποιο ε, λογικό χρόνο. Η Άννα Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω τη μετρική μου γλώσσα. Ευχαριστώ, Κόνη. Πραγματικά χαίρομαι που σε βλέπω εδώ. Επιτέλους, επιτέλους θα μιλήσουμε για τα πλοία. Εφόσον έχουμε επανεξετάσει όλα τα μέσα μεταφοράς. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που επιτέλους ε, συζητούμε και αυτό το θέμα. Και ο Πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει υπερβολικό δυναμικό σε ό,τι αφορά τα παλιά πλοία, όμως οι περισσότεροι ε, πλειοκτήτες γνωρίζουν πολύ καλά ότι όταν πρέπει να αγοράσουν νέα πλοία, πρέπει να λάβουν υπόψη ότι θέλουμε μηδενικές εκπομπές. Γιατί είναι λιγότερο ακριβό για εκείνους, είναι πιο φθηνό για εκείνους να το εξετάσουν μακροπρόθεσμα το θέμα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα πλοία για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όταν μιλώ λοιπόν με τους ε, Δανείους εφοπλιστές ε, γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και ελπίζουν σε διεθνές επίπεδο να καταφέρουμε να απευθυνθούμε σε ε, περισσότερους φορείς από ό,τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Γνωρίζουν επίσης ότι μεγάλες επιχειρήσεις στρέφονται προς ε, νέες μορφές καυσίμων, όπως τα βιοκαύσιμα. Πράγματι λοιπόν, ήδη υπάρχουν εξελίξεις ε, στον κλάδο και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερως. Θα ήθελα όμως να θέσω το εξής ερώτημα. Πώς μπορούμε να έχουμε ελπίδες παρακολούθησης ε, των εκπομπών σε ό,τι αφορά όλους αυτούς τους ρήπους, όλα αυτά τα αέρια του θερμοκηπίου. Γιατί ταυτόχρονα Μιλάμε για όλα τα είδη πλοίων, τα αλληλευτικά, τα πλοία εμπορευματο... <laughs> εμπορευματοκιβωτίων. Αλλά και ε, πλοία που εξυπηρετούν ε, ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές, όπως Ακτική, Ανταρκτική. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς μπορούμε να επιβλέψουμε αυτή τη μείωση με πολύ απλό και απτό τρόπο. Και κάτι ακόμα. Υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ πλειοκτήτων και μεταξύ των αυλωτών. Τους εφοπλιστές μπορούμε να τους ρυθμίσουμε, αλλά τι κάνουμε με τους ναυλωτές. Εκείνοι δεν έχουν απολύτως καμία υποχρέωση. Πρέπει κάτι να γίνει και με αυτούς λοιπόν, με τους ναυλωτές. Και πολύ σύντομα θα ήθελα να ε, πω δύο λόγια για την ε, διάσκεψη για το κλίμα. Και εγώ έχω ένα μικρό ερώτημα. Με τα όσα είπε και ο προλαλής για το send more money, πώς θα στείλουμε περισσότερα χρήματα. Ξέρω ότι στην Ευρώπη μας βλέπουν μάλλον ε, απ' έξω σαν τους πλούσιους, αλλά αυτή η ιδέα του send more money μου φαίνεται επικίνδυνη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην χάσουμε τη στήριξη των Ευρωπαίων που δεν μπορούν να στηρίξουν μια τέτοια προσέγγιση του send more money. Πώς θα δράσουμε λοιπόν με διαφορετικό τρόπο για να διασφαλίσουμε ότι θα στηρίζουμε τους υπολείπους, αλλά όχι με οικονομικούς πόρους θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα διαφορετικό τύπου καρότο για να δώσουμε κίνητρα στους άλλους να συνεργαστούν, όχι με ε, κίνητρα χρηματοδότησης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιμάντσικη. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα προσεκτικά τα όσα είπατε για τη διασκέψη στη Βαρσοβία. Ο κύριος Πρόεδρος ε, είπε ότι υπερβήκαμε τις προσδοκίες και εσείς είπατε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα. Πολλοί απογοητεύτηκαν, αλλά αυτό δεν μας εκπλήσει. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τα παγκόσμια δεδομένα, τα πραγματικά δεδομένα και έτσι δεν μπορούμε να μιλάμε για έκπληξη. Μιλάμε για μια παγκόσμια συμφωνία και αλλαγή της γλώσσας, της διατύπωσης, αλλά αυτά δεν αλλάζουν πολλά. Οπότε με εκπλήσει ότι τα λέμε αυτά. Δεν υπάρχει καμιά ε, ξαφνική ρήξη και έλευθη λύση στον ορίζοντα. Θέλω να πιστέψω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε ως Ευρώπη, αλλά αυτή η πολιτική του να αποτελούμε υπόδειγμα υπάρχει μια διαφορά μεταξύ εμάς και του υπόλοιπου κόσμου. Ό,τι κάνουμε εδώ είναι πολύ ακριβές. Έχουμε κάποιες διενέξεις μεν, αλλά άλλες χώρες όπως η Κίνα δεν ακολουθούν, δεν εισάγουν αλλαγές. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Όσον αφορά το χάλιβα, τα προϊόντα χάλιβα, έχουμε έχουμε δασμούς αντι-dumping σε ύψος 70%. Και έχουμε και αυτό το περιβάλλον κρίσης ε, το οποίο βιώνουμε και θα συμφωνήσω με τον Έλληνα συνάδελφο. Συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές. Έχουμε το θέμα της ε, ένδυας ε, έλλειψης καυσίμων στις χώρες μας, στην Πολωνία σε ορισμένα νοικοκυριά. Το 40-50% των δαπανών του νοικοκυριού πηγαίνει στην ενέργεια. Δεν αναφέραμε σε αυτά μόνο γιατί έχουμε εκλογέ του χρόνου. Πρόκειται για αδιάστατα γεγονότα, ρεαλιστικά, πραγματικά γεγονότα και πολλοί κόσμοι αναρωτιέται γιατί πρέπει να δεχθούμε νέες μειώσει, νέους στόχου, ε, και να διαλέξουμε νέους δείκτες. Για παράδειγμα, ε, ε, αριθμούς τόνους άνθρακα, διεξουδίου του άνθρακα κατά κεφαλήν. Πρέπει να δούμε καθαρά αυτές τις διαφορές ε, τις χώρες που, κάνουν, που είναι διαφορετικές στην Πορτογαλία, στην Πολωνία, στην Ελλάδα έχουμε εισαγεί πολλές μειώσεις σε σχέση με το σημείο από όπου ξεκινήσαμε οι εκπομπές μας ε, κατά κεφαλή είναι χαμηλότερες από τη Γερμανία και πολύ συχνά αναφέρονται σε εμά ω ε, του σημαντικού ρεπαντέ τη Ευρώπη. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σα στο γεγονό ότι η μεγαλύτερη προσδοκία αυτή τη στιγμή είναι ότι χωρίς αυτή την παγκόσμια συμφωνία το μέλλον του πλανήτη μας είναι αμφισβητήσιμο. Η συμβολή της Ευρώπης μειώνεται λόγω της κρίσης. Ε, άλλοι είναι πιο γρήγοροι από εμάς και εμείς δεν καταφέρουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Σε αυτό το περιβάλλον παγκόσμιου συναγωνισμού εμείς δεν βρισκόμαστε στην πρώτη θέση και είναι πολύ σημαντικό. Η οικονομία μας δεν είναι ανταγωνιστική παγκόσμια, είμαστε ανταγωνιστικοί στο κλίμα, αλλά και αυτά μας τα λένε οι πολίτες μας. Και εμείς ε, ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή ασφάλεια και τους πολίτες μας. Στη συνθήκη της Λεσσαμόνας αναφέρεται σαφώς ότι όλες μας οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν πρέπει να επηρεάζουν το ενεργειακό μείγμα των επιμέρους κρατών μελών και την ενεργειακή του ασφάλεια. Αναφέρομαι όλα αυτά, διότι ε, λεπτομερής ανάλυση σε κάθε κράτος μέλος ε, αλλάζει τη συζήτηση περί εκπομπών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους πολίτες μας. Ε, δεν μπορούμε να τους αφήνουμε στην άκρη. Ελπίζω ότι η Επιτροπή δεν πρόκειται να λάβει αποφάσεις χωρίς να λάβει υπόψη τη τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου Έχουμε σημαντικά αρχή αυτή τη στιγμή. Έχουμε τον κύριο, την εκθέση του κ. Σμάνσκι, την οποία μελετάμε αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω ότι όλες αυτές οι σκέψεις μετά από τη Βαρσοβία θα πρέπει να μας αναγκάσουν να εξετάσουμε λεπτομέρως, να λάβουμε υπόψη λεπτομέρως όλους αυτούς τους παράγοντες. Δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι. Πιστεύω ότι οι στόχοι αυτοί είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε συναγωνισμό με τον κόσμο. Καρλ Χάιντ Φλόρεντ, παρακαλώ. Άφωνο έχει μείνει ο κύριο ε, Φλόρεντ, λέει ο κύριο Γκρότ. Θα πει τίποτα, Καρλ Χάιντ. Οκ. Περιμένουμε. Και μετά Γεμπράντι. Α, δεν είναι παρόν ο Γεμπράντι. Α, ούτε άλλος. Α, ωραία, δεν θα μιλήσει ούτε ο κύριος Φλόρεντς. Λοιπόν, κάτι ζήτησε, για κάτι ζήτησε ε, το λόγο πάλι η κυρία Μακάβεν και μετά η κυρία Σούζα. Νομίζω ότι θα συζητάγαμε κατόπιν την έκθεση για τις ναυτιλιακές εκπομπές. Επειδή είναι, λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, έχουμε συγχωνεύσει τις δύο συζητήσεις. Δεν θα κάνουμε άλλη συζήτηση. Κατόπιν, λέει ο πρόεδρος, κατόπιν θα γίνει άλλη συζήτηση. Α, οπότε δεν χρειάζεται να πάρω το λόγο τώρα, λέει κύριε Μακάβαν. Πολύ ωραία. Ωραία, λέει ο πρόεδρος. Σούζα. Pa samo bih se kratko htjela zahvaliti povjerenici na ovom izvješću nakon e, Varšave. svakom slučaju... Επιτρέψτε μου να αρχικά να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο για την ενημέρωση που μας παρουσίασε όσον αφορά τη διασκέψη στη Βαρσοβία. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που όλα τα θεσμικά όργανα και ειδικά η Επιτροπή Περιφερειών ασχολούνται με το θέμα. Έχουν πολλά να πούν αυτοί, η Επιτροπή Περιφερειών, γιατί βρίσκονται τόσο κοντά στους πολίτες. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία. Είπαμε ότι υπάρχουν πολλοί κανόνες ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και είπαμε ότι αποσκοπούσαμε σε μια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Αλλά ήθελα πρώτα απ' όλα να μιλήσω για κάτι άλλο. Για το γεγονός ότι έχουμε όλο και περισσότερα και μεγαλύτερα κρουαζιερόπλαια. Πρόκειται για μια ανθυρή βιομηχανία, ένα ανθυρό τομέα Έρχομαι από το, τώρα από το Ντουμπρόβνικ ε, όπου εδώ και 5-6 χρόνια στο λιμάνι της πόλης βλέπουμε τεράστια κρουαζιερόπλια. Το Ντουμπρόβνικ ε, αποτελεί, ανήκει στην παγκόσμια κληρονομιά και προστατεύεται αντίστοιχα. Οι εκπομπές ρήπων από τα κρουαζιερόπλια είναι τεράστιες. Γι' αυτό το λόγο με ενδιαφέρει τόσο πολύ το ζήτημα αυτό. Μιλήσαμε για τη διαχείριση των θαλασσίων αγαθών, την ολοκληρωμένη διαχείριση. Εμείς θα θέλαμε εδώ να έχουμε μια ολοκληρωμένη διαχείριση, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι η Αδριατική δεν αποτελεί όλη κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι κάποιες χώρες γύρω από την Αδριατική δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπόκειται λοιπόν στους ίδιους κανόνες. Ε, υπάρχει το θέμα της Τουρκίας και των πλοίων στα δρομολόγια μεταξύ Ελλάδα και Τουρκίας. Πώς μπορούμε να υποβα... επιβάλλουμε τους ίδιους κανόνες σε όλα αυτά τα σκάφη, σε όλα αυτά τα πλοία. Συνεπώς είμαι υπέρ της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Επίσης, με ποιο τρόπο μπορούμε να δώσουμε κίνητρα στις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου στις θαλάσσιες μεταφορές. Επίσης ε, υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία οι χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ακολουθήσουν. Ε, ε, εάν υπάρξουν τέτοια μέτρα, τι επιπτώσεις θα έχουν. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτησή μας και η Επίτροπος τώρα θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι κατάλαβα, μετά από αυτή τη συζήτηση ε, θα υπάρξει και πιο συγκεκριμένη συζήτηση και υπάρχει και ομάδα υπερογνωμόνων της Κομισιόν που θα μείνει εδώ και να απαντήσει σε τέτοια πιο ειδικά ερωτήματα. Προς τον κύριο Ζήμπερ, να ξεκαθαρίσω, γιατί κατανοώ ότι δική σας επιφύλαξη και ανησυχία λέτε ότι δεν πρέπει να έχουμε στόχους, δεν πρέπει να έχουμε το ένα, το άλλο και το καθεξής. Ούτε αυτό έχουμε εδώ. εφόσον μιλάμε για σταδιακή προσέγγιση, αυτό είναι το πρώτο στάδιο, το πρώτο βήμα. Ό,τι είδου σύστημα για να επιλέξουμε ή επιθυμούμε, όποιο σύστημα από αυτά που ανέφερε ο κύριος Σκυλακάκης, ε, πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα MRV. Γι' αυτό και δεν προδικάζουμε τι είδους σύστημα θα είναι αυτό, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Όμως έχουμε ε, το υπέδαφος, αυτό το υπόβαθρο που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε κάποια στιγμή με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Γι' αυτό και βασιζόμαστε σε εκτενείς διαβουλεύσεις και με τον κλάδο. Και ο κύριος Κάλλας και εγώ είχαμε τρεις συνεδριάσεις υψηλού επίπεδου. Οι εμπειρογνώμονες μας είχαν ακόμα περισσότερες τέτοιες συναντήσεις με όλες ε, τις πλευρές ε, του κλάδου, με όλα τα διαφορετικά μέρη. Και η δική μου εντύπωση είναι ότι αυτό που προτείνουμε εδώ το MRV, είναι κάτι το οποίο δεν είναι αμφιλεγόμενο. Όλοι θεωρούν ότι όπως και να έχει είναι ένας λογικός τρόπος ε, να προχωρήσουμε, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε επίπεδο IMO. Επομένω, περί αυτού πρόκειται. Δεν μιλάμε πλέον για συγκεκριμένους ε, στόχους. Είναι το πρώτο βήμα. Νομίζω ότι έτσι απαντώ και σε κάποιες από τις ε, Παρατηρήσει του κυρίου Σκυλακάκη για την τιμολόγηση, κατά πόσο πρέπει να είναι αγορακεντρικός ε, μηχανισμός ε, ή κάποιο τέλος, φόρος. Αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στον IMO και βεβαίως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι μέλος του IMO, όμως υπενθυμίζω ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει και συνιστώ μάλλον να συνεργαστούν και να προωθήσουν αυτό το σημείο και είναι θετική εξέλιξη ότι και η Αμερικανική πλευρά έρχεται με συγκεκριμένε προτάσεις. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες πιθανότητες, καλές πιθανότητες να κάνει αυτό το βήμα ο IMO, όμως βεβαίως με τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ασκήσουν πιέσεις για να γίνει αυτό. Είπατε ότι θα πρέπει να έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται με το αμερικανικό σχέδιο. Ήδη αυτό κάνουμε. Είπατε επίσης ότι θα πρέπει ε, να προσπαθήσουμε να θεσπιστεί ένα παγκόσμιο σύστημα. Ακριβώς αυτό θέλουμε και εμείς να επιτύχουμε. Μας ρωτήσατε πώς μπορούμε να έχουμε μια ιδέα των ε, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Βασιζόμαστε στην κατανάλωση καυσίμων και θα υπάρχουν δεδομένα πάνω σε αυτό. Γι' αυτό και θέλουμε το σύστημα να είναι όσο δυνατόν απλούστερο για να μην ε, αναγκαστούμε ε, να βρούμε νέε διοικητικέ διαδικασίες με νέο διοικητικό άχθος. Θα βασιστούμε όσο μπορούμε σε αυτά που ήδη υπάρχουν. Αλλά μετά υπάρχει και αυτή η συζήτηση για τα μεγάλα και τα μικρότερα πλοία. Είναι σαφές ότι όσο μικρότερα πλοία συμπεριλάβουμε, τόσο υπάρχει κίνδυνο κίνδυνος αυξημένου διοικητικού άχθους. Τώρα, τι συμβαίνει με τον αυλωτή. Το ανέφερα και προηγουμένω. Δεν θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα με αυτό το συγκεκριμένο μέτρο, γιατί αφορά άλλο ζήτημα. Όμως υπάρχει θετική εμπειρία στον κλάδο. Ο μεγαλύτερος δανός εμπορευόμενος ε, ακολουθεί κάποιες ευέλτιστες πρακτικές. Υπάρχουν τέλος πάντων τέτοιες πρακτικές που θα είναι ενδιαφέρουσες και για τους ναυλωτές. Όμως το θέμα είναι ποιος θα έχει το κίνητρο για να κάνει κάτι εδώ. Και για να είμαι σαφής, εδώ δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση προς οποιονδήποτε σε αυτή την πρόταση. Και τέλος, κύριε Σούσα, για ε, τα κουραζιερόπλια. Ναι, πράγματι είναι περίπλοκο ε, αυτό το ζήτημα με τα ε, οξύδια ζώου του θείου και το καθεξής. και είπατε μπορούμε κάπως ε, να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, αναφερθήκατε συγκεκριμένα στην Αδριατική. Νομίζω ότι υπάρχει ένα καλό πρότυπο ε, αν ακολουθήσουμε τις ρυθμίσεις που είχαμε στη Βαλτική. Εκεί προσπαθήσαμε να επιλύσουμε το ζήτημα τοπικά με τους ε, άλλους εταίρους, με τρίτες χώρες ακόμα. Για τις διαπραγματεύσεις Ευχαριστώ τον Ρίτσαρντ Σέιμπερ που είπε ότι θα συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Εδώ χρειαζόμαστε και τις κυβερνήσεις, ε, τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, τους Ευρωβουλευτές, γιατί συμφωνώ ότι είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Και τον ανέφερα εν συντομία και στην αρχή. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε ανοιχτά για τα προβλήματα. Στη Βαρσοβία είχα την αίσθηση ότι όλοι οι φίλοι μας ε, και στις αναπτυσσόμενες χώρες, ε, στις αφρικανικές χώρες, στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής Αμερικής θέλουν να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση με εμά. θέλουν φιλοδοξία σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Όμως, για να είμαι ειλικρινής, ε, μας δημιουργεί ένας προβληματισμός. Ε, αυτή η ομάδα ε, που σπατάλησε πολλές ώρες για να δει αν μπορούμε να αποκαταστήσουμε τις υφιστάμενες εκπομπές στο παράρτημα 1. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για την ευρωπαϊκή πλευρά, αλλά για όλε τι πλευρέ που θέλουν να υπάρξει κατάλληλη επίλυση του προβλήματο για το κλίμα, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν κρατήσουμε αυτή την παλιά γραμμή. Γι' αυτό αναφέρθηκε συνάδελφο προηγουμένω και στη χρηματοδότηση. Βεβαίω και θα πρέπει να βοηθήσουμε τι λιγότερο αναπτυγμένε και περισσότερο ευάλωτε χώρε στον κόσμο να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να ακολουθήσουν τον δρόμο τη ε, ε, βιώσιμη ανάπτυξη. πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε τη δημόσια χρηματοδότηση για το περιβάλλον για να υπάρξει μόχλευση ε, από τον ιδιωτικό κλάδο για επενδύσεις ε, και ούτω καθεξής. Όμως, σε κάποιες από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες στην ομάδα των αναπτυσσόμενων χωρών, βεβαίως και δεν μπορούμε να μιλούμε για χρηματοδότηση. Θα πρέπει να συμβάλλουν και θα πρέπει να αναλάβουν τις δεσμεύσεις τους. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι και ελπίζω και εγώ να μην χρειαστεί να δαπανίσουμε πολύ χρόνο μέχρι το Παρίσι για να επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά τις ίδιες συζητήσεις κατά πώς θα πρέπει να υπάρξει αυτό το ε, τείχος προστασίας ή όχι. Δεν χρειαζόμαστε νέα τείχη πρέπει να διαμορφώσουμε τον, το νέο μελλοντικό καθεστώς όπου θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε. Βεβαίως, όχι όλοι εξίσου, κάποιοι θα πρέπει να συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλους. Και θα πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση. Όμως, η διάκριση δεν μπορεί να ε, γίνεται μεταξύ των μελών των 92 και των υπολείπων. Για την ε, κυρία Μακάβεν. Αναφερθήκατε σε αυτό το κόστος ε, για το 2030 και πόσο γεννούμαστε σε ό,τι αφορά το εγχείρημα το 2030 από πλευρά Κομισιόν. Η εξολόγηση αντικτύπου που προετοιμάζουμε βεβαίως και αναφέρεται ε, στον αριθμό των στόχων, την ε, αλληλεπίδραση μεταξύ των στόχων και το επίπεδο φιλοδοξιών. Αλλά βεβαίως θα θίξουμε και το ζήτημα του κόστους, θα υπάρξει ανάλυση του ενεργειακού κόστους θα ληφθεί υπόψη και το σκέλος της απασχόλησης όταν έχουμε αποδοτικότητα και ανανεώσουμε σε πηγές ενέργειας, ε, δημιουργούμε περισσότερες θέσεις εργασίας. Όμως βεβαίως και θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την κλιματική αλλαγή για να ε, προκαλούμε την καινοτομία, τις εξαγωγές, την απασχόληση. Η ενεργειακή εξάρτηση θα είναι άλλο ε, σκέλος. Η Ευρώπη την είναι, αυξάνει την εξάρτησή της. 545 δις πληρώσαμε πέρσι ως Ευρώπη για την εισαγωγή ορεικτών καυσίμων. Χρήματα τα οποία πήγαν προς τα έξω, στο εξωτερικό, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Κατάρ, Σαουδική Αραβία και το καθεξής, αντί να τα επενδύσουμε στην ε, Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία, στην Πολωνία, οπουδήποτε αλλού. Και αυτό λοιπόν είναι τμήμα του προπαρασκευαστικού έργου αυτού. Τέλος, για τις επιδοτήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και εδώ εξετάζουμε πώς μπορεί να γίνει αυτό με οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο. Όσοι θέλουμε να συνεχιστεί η ανάπτυξη των ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα πρέπει να μας απασχολήσει το πώς θα αποφύγουμε την υπερστήριξη των ανανεώσιμων. Γιατί μέχρι το 2020 κάποιες από αυτές τις τεχνολογίες θα είναι πιο όριμες, βεβαίω δεν θα πρέπει να επιδοτούνται. Πώς θα βρούμε λοιπόν έναν πιο ευέλικτο και δυναμικό τρόπο επιδοτήσεων. Όλα αυτά τα στοιχεία θα συμπεριλαμβάνονται. Βεβαίω πρέπει να πω ότι ένα από τα στοιχεία τα οποία θα προσπαθήσω εγώ να επιτύχω μέσω αυτού του εγχειρήματο είναι να ξεκαθαρίσουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει αυτή η συζήτηση ότι το μέσο νοικοκυριό θα έχει αύξηση 112 λιρών στον λογαριασμό τους στις δαπάνες τους για την ενέργεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κονδύλιο αν κάποιος βρίσκεται στο Μάντσεστερ. Όμως αυτό συνδέεται με την ε, κλιματική πολιτική και ούτω καθεξής. Η, το, το κόστος των ενεργειακών υποδομών, του κλίματος και η ε, τιμές του, του χονδρικού εμπορίου μπορούν να αιτιολογήσουν τα 35, τις 35 λίρες από τις 112. Υπάρχει λοιπόν μετά και ένα πολύ σημαντικό χάσμα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι ακριβώς ισχύει στην όλη αυτή τη συζήτηση. Και τέλος, πρέπει να έχουμε πολύ οικονομικά αποδοτικό ενεργειακό σύστημα στην Ευρώπη. Πολύ οικονομικά αποδοτικές ενεργειακές πολιτικές θα πρέπει να έχουμε στην Ευρώπη. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτό. Αλλά να πω ξεκάθαρα ότι αν υπάρχει μόνο μία παράμετρος ότι χρειαζόμαστε τη φθηνότερη δυνατή ενέργεια, τότε ξέρουμε τι θα πάρουμε. Περισσότερο άνθρακα. Δεν είναι δύσκολο. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Και βεβαίως μετά δεν μπορούμε να έχουμε μία εύλογη περιβαλλοντική πολιτική. Στην ανακοίνωση την οποία ανέφερε και ο Ρίτσαρτ, θα πρέπει να είμαστε σαφείς ότι δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη ε, μετάβαση στην οικονομία χαμηλού άνθρακα χωρίς κανένα κόστος. Υπάρχει κόστος, όμως μακροπρόθεσμα υπάρχουν ε, παράλληλα ωφέλη. Αυτή είναι η δυσκολία. Ε, είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε βεβαίω στου υπόλοιπου φορεί. Και τέλο για τον κύριο Σουμάνσκι αναφέρατε όσους έχουν ήδη καταβάλει προσπάθειες. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όταν μιλούμε για δείκτες, κριτήρια, ότι πρέπει να αξιολογήσουμε τι είναι δίκαιο και τι όχι. Βεβαίω το μελλοντικό σύστημα καθεστώ δεν θα πρέπει να τιμωρηθείτε αν ήσασταν από του πρώτου που έκαναν τη μετάβαση. Βεβαίω θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το στοιχείο. Σε διεθνέ επίπεδο όμω θέλουμε όλοι μας, ακόμα και όσοι έχουν κάνει πολλά, να αναγκαστούμε να κάνουμε περισσότερα για να μείνουμε στους δύο βαθμούς. Το πρόβλημα και το, η μεγάλη συζήτηση είναι πώς ε, ακριβώς θα εμπλέξουμε όλους τους φορείς σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Κόνη Χέντεγκαρντ, για αυτήν την αναλυτική απάντηση στα ερωτήματα που είχαν τεθεί και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία για τις επόμενες εβδομάδες ε, στην πορεία προς το Παρίσι. Πρέπει να υπάρξει επιτυχία, πρέπει να επιτύχουμε ορισμένα πράγματα, ουσιώδη αποτελέσματα για ένα καλύτερο μέλλον, για το κλίμα, αλλά και για την οικονομική κατάσταση. Γιατί αυτά τα δύο είναι συνδεδεμένα, πολύ στενά συνδεδεμένα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Οπότε, οπότε πάλι στα δικά μας θέματα τώρα τα καθημερινά, την γενικότερη συζήτηση την κάναμε. Έκθεση λοιπόν του συναδέλφου Σκύλα Κάκη που ασχολείται ακριβώς με αυτά που τώρα μόλις συζητούσαμε, δηλαδή τι θέλουμε να κάνουμε στον ναυτιλιακό τομέα. Έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα να δώσω το λόγο στον εισηγητή για να μας προσθέσει το θέμα. Παρακαλώ, ο κύριος Κυλακάκης. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί είπα τα περισσότερα στην προηγούμενη μου παρέμβαση. Απλά έχω λίγα πράγματα να προσθέσω. Πιστεύω ωφέλιμα. Τη γενική εισαγωγή την έκανα ήδη. Ας περάσουμε σε κάποιες λεπτομέρειες. Η πρώτη έχει να κάνει με το είδος των στοιχείων που θα δημοσιεύουμε. Εγώ προτείνω να δημοσιεύουμε όλα τα στοιχεία αλλά ανώνυμα όσον αφορά το όνομα του πλοίου και της εταιρείας. Έτσι θα παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για ζητήματα απόδοσης που θέλει να γνωρίζει η Κομισιόν αλλά θα μας γλιτώσει από πολλές παραπλανητικές συζητήσεις που θα μπορούσαν να πλήξουν την όλη διαδικασία γιατί πρέπει κανείς να αντιληφθεί ότι η ενεργειακή απόδοση ενός πλοίου είναι περίπλοκο ζήτημα δεν ορίζεται μόνο βάση του καυσίμου ή του φορτίου. Επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, από τα θαλάσσια ρεύματα, από το χρόνο που έχει παρέλθει από τη στιγμή που ένα πλοίο μπήκε σε dry dock. Μπορεί ένα πλοίο να είναι πιο ενεργειακά αποδοτικό μόλις αυτό βγήκε από τον dry όπου έχει καθαριστεί το κήτος και η προπέλα και να μειωθεί η ενεργειακή του απόδοση ε, με τον καιρό και να βρεθεί στα χαμηλότερα σημεία πριν ξαναμπεί σε dry dock για καθαρισμό. Ε, επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πολλές φορές είναι σημαντική η απόδοση ως προς τις αγορές. Ε, για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα δρομολόγιο από τη Γαλλία προς την Αλγερία. πηγαίνει το πλοίο γεμάτο διότι η Αλγερία εισάγει πολλά πράγματα και γυρίζει το πλοίο άδειο διότι εξάγει τα κάψιμα η Αλγερία μέσω αγωγών. Ποια είναι η ενεργειακή απόδοση σε αυτό το ταξίδι, για παράδειγμα. Άλλε φορέ πρέπει να πάει ένα πλοίο πολύ γρήγορα για να παραλάβει ένα εμπόρευμα και τέλο υπάρχουν πολλέ τέτοιε διαφορετικέ περιπτώσει. Τι ενεργειακή απόδοση θα μετρηθεί, μάζα ή βάρος διότι είναι εντελώς διαφορετική η ενεργειακή απόδοση αν ένα πλοίο είναι βαρύ. Αλλά υπάρχουν, πλοία που, υπάρχουν φορτία που ε, καταλαμβάνουν πολύ χώρο, ε, ε, τα πλοία γενικώ καταλαμβάνουν πολύ χώρο, αλλά μπορεί να μην είναι βαριά αναλόγω με το φορτίο. Γι' αυτό τον λόγο οι Αμερικανοί στον IMO έχουν υποβαλεί τρεις διαδοχικές προτάσεις. Τη μία χωρίς ε, έργο μεταφοράς, τη δεύτερη με έργο μεταφοράς και η τρίτη βασίζεται με το χρόνο στη θάλασσα. Εγώ προτείνω να μετράμε βάση του χρόνου στη θάλασσα. Είναι σημαντικό διότι μπορούμε να βασιστούμε στα στοιχεία του χρόνου στη θάλασσα. Το φορτίο το να λάβουμε το φορτίο υπόψη ως παράγοντα πιστεύω δεν θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε ό,τι καλύτερο για την ενεργειακή απόδοση των πλοίων. Τέλος, δεν θέλω να επεκταθώ υπερβολικά σε λεπτομέρειες, θέλω να ακούσω και τα όσα έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος πιστεύω ότι τα οξύδια του αζότου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Δεν είναι κάτι εύκολο στη μέτρηση. Συνεπώ πρέπει να συζητήσουμε πώ θα γίνει. Αλλά σύμφωνα με αυτή τη μελέτη που σα ανέφερα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντο, τα οξύδια του αζότου έχουν και αρνητικέ και θετικέ επιπτώσει, τόσο σημαντικέ όσο το διοξίδιο του άνθρακα αλλά με μεταβλητούς παράγοντες που οδηγούν σε πολύ μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Επίσης τα οξύδια του αζότου σχετίζονται άμεσα, συνδέονται άμεσα με τον τρόπο κατασκευής των μηχανών. Μπορεί να έχουν κατασκευαστεί μηχανές για ε, περισσότερα οξύδια του αζότου και λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα και αντίστροφα. Λόγω της αβεβαιότητας λοιπόν αυτής Δηλαδή υπάρχει και η θετική πλευρά του ε, οξυδίου του αζότου ότι μειώνει το μεθάνιο. Ε, πιστεύω ότι είναι σημαντική λοιπόν η μέτρηση των οξυδίων του αζότου. Και αντίστροφα με τα αέρια ε, οξυδίου του θείου, τα ε, οξύδια του αζότου θα αυξηθούν στο μέλλον. Οπότε πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεν πρότεινα το μαύρο άνθρακα για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Δεν είναι τόσο σημαντικός στην παρούσα φάση ως ε, ρήπος. Προτείνω λοιπόν να επεκτείνουμε το παιδί εφαρμογή από το διοξίδιο του άνθρακα και στα οξύδια του αζότου. αλλά όχι στους υπόλοιπους ρήπους, διότι αυτοί είναι οι δύο βασικοί παράγοντες που κατά την απόψη μου ε, έχουν, έχει νόημα να λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Οι εκπρόσωποι τώρα των ε, πολιτικών ομάδων. Πρώτη η Λίντα. Στούτα μετά και μετά η Άννα Ρόσμπαχ. Η Λίντα. Δεν είναι κανείς από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Ο κ. Αρσένης ε, ζητεί συγγνώμη που δεν παρευρίσκεται σήμερα, δεν είναι καλά σήμερα. Μου ζήτησε όμως να μεταφέρω τις σκέψεις του επί της πρότασης. Πρώτον, Άκουσα τα όσα αναφέρθηκαν ε, από την Κομισιόν για τον εξοπλισμό για τα νόξ, για τα οξύδια του αζότου. Ο Κρήτον όμως λέει ότι χαιρετίζει την ε, πρόθεση της Επιτροπής να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή ε, και στα νόξ. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε ευρύτερο πεδίο εφαρμογή για να καλύπτουμε εκπομπέ και πέραν του διευθυντήτου του άνθρακα. Είναι επικρατικό σε ό,τι αφορά την διαγραφή του εμπορεύματος ε, που ε, μεταφέρεται από τον κατάλογο των ε, στοιχείων που θα πρέπει να παρακολουθούνται. Γιατί έτσι υπονομεύεται ο στόχος της διευκόλυνσης δευτερογενούς αγοράς στα πλοία. Τώρα, για το κατά πόσο πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα, να επενθυμίσουμε ότι τμήμα του κλάδου της βιομηχανίας συμφωνεί με την προσθήκη τα περισσότερα από αυτά τα δεδομένα είναι ήδη διαθέσιμα, παράδειγμα για τις προλογικές δηλώσεις. Σε ό,τι αφορά τι μεθόδου παρακολούθηση για τον υπολογισμό τη ε, πραγματική κατανάλωση καυσίμων, να υπογραμμίσουμε ότι δεν είναι όλα αυτά τα στοιχεία εξίσου ακριβή. Θα πρέπει να κινηθούμε βαθμιδών και να επιλέγουμε πάντα τι πιο αποδοτικέ και ε, ακριβεί ε, μεθόδου. Συμφωνούμε με τι εξουσιοδοτήσει που δίνονται στην Κομισιόν θα πρέπει τα συστήματα MRV της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ευθυγραμμιστούν με τα διεθνή πρότυπα και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει κάτι εξοδότηση πράξη. Ε, το, το, το, αντίστοιχο πρόβλημα έχουμε και εμείς, οι σκιώδεις ε, είναι άρρωστη, όμως ε, θα ήθελα να πω δύο λόγια εκ μέρους της. Και εκείνη χαιρετίζει το γεγονό ότι έχετε μειώσει το κατόφλι τη χωρητικότητα και έχετε συμπεριλάβει τα οξύδια του αζότου. Αυτό κινείται προ την κατεύθυνση. Ωστόσο, θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετό το να έχουμε μόνο ε, την παρακολούθηση υποβολή εκθέσεων και ταυτοποίηση. Είναι καλή, καλό πρώτο βήμα, όμως θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο σύστημα ETS όπως ψήφισε το Κοινοβούλιο το 2008 και από τότε συμφωνήσαμε ότι αν ο IMO μέχρι το 2011 δεν το έχει θεσπίσει θα το εισαγάγουμε εμείς. Εμείς ε, εμένουμε λοιπόν σε αυτό το στοιχείο, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον κανονισμό. Και σε περίπτωση που το Συμβούλιο δεν είναι διατεθειμένο να το κάνει τώρα, θα πρέπει να ε, προβλέψουμε ένα πολύ αυστηρόχρονο διάγραμμα για την Κομισιόν. Γιατί ήδη αυτό υπήρχε σε αιτιολογική σκέψη ε, στο πακέτο για το κλίμα του Συμβουλίου. Ε, είμαι αλλεργικό ε, στα εμπιστευτικά δεδομένα, επομένω η τροπολογία 59 για μένα δεν, ε, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Πάντα η εμπιστευτικότητα θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση και μόνο όταν αυτό είναι απολύτω απαραίτητο οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων βεβαίως ε, θα πρέπει να ε, διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο, το ώστε να μην έχουμε τις εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες. Όμως θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ε, να γίνεται αυτή η υποβολή εκθέσεων. Κατά τα λοιπά, σας ευχαριστώ και προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία σε ό,τι αφορά τους συμβιβασμού. Ευχαριστώ, Ανά Ροσπαχ. Ευχαριστώ. Υπάρχει το ζήτημα των αξιδιών του αζότου, το οποίο με απασχολεί. Ο σχεδόν ο Μάρτιν Κάλαραν, δεν ε, κατάφερε να παρευρεθεί σήμερα. Έχει διαφορετική θέση από μένα σε προσωπικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τα αξιωδία του ζώου Θα σας διαβάσω λοιπόν τη δική του τοποθέτηση. Η Κομισιόν πρότεινε ο κανονισμός να συμπεριλάβει και τα πλοία ε, των χωρητικότητας 500 ε, τόνων. Όμως 5.000 ε, τόνων, συγγνώμη, αλλά δεν θεωρούμε ότι είναι κατάλληλο να περάσουμε στους 400 τόνους συνολικής χωρητικότητας. Αυτό δεν είναι πρακτικό για τους ιδιοκτήτες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι μεγάλος αριθμός χωρών, το πλοίων, συγγνώμη, έχει ήδη περιορίσει τις εκπομπές τους πρέπει να υπάρχουν και άλλες ε, ρήτρε ε, ε, στη νομοθεσία ανέφερε ο εισηγητής και εγώ συμφωνώ. Βεβαίω πράγματι θα υπάρξει ένα αυξημένο διοικητικό άκθος και για τις αρχές, τις εθνικές αρχές που θα πρέπει να τα ελέγχουν όλα αυτά. Έτσι αυξάνονται και οι πιθανότητες απάτης λόγω της έλλειψης ελέγχων και και παραβιάσουν γενικότερα των κανόνων. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει πολύ ε, σημαντική αύξηση του διοικητικού άχθους, ιδιαίτερα για τα πλοία που κάνουν σύντομα δρομολόγια, για παράδειγμα για τα ferry boat. Και υπάρχει και το εξή στοιχείο το οποίο θα πρέπει να παρακολουθούμε. Υπάρχει όλος αυτός ο μεγάλος αριθμός των ε, ferry boat. Θα πρέπει να δούμε μήπως μπορούμε να βρούμε διαφορετικά ειδικό τύπο μέτρων και όχι μέτρο αναδρομολόγιο. Θα μείνω εδώ. Οπότε να δώσω τώρα το λόγο στην ε, Επιτροπή και μετά πάλι ο εισηγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και όλους όσους ε, σχολίασαν την πρόταση και το σχέδιο έκθεση, έκθεσης του εισηγητή. στόχος με την πρότασή μας είναι να συμβαδίζει με τις διεθνείς διαδικασίες. Αυτό το υπογράμμισε και η Επίτροπος. Η προσέγγιση λοιπόν αυτή είναι και μετριοπαθής και επικοδομητική αλλά βασίζεται στις βασικές αρχές και στόχους της ενωσιακής πολιτικής. Σχόλια τώρα και παρατηρήσεις Πρώτον, τι πληροφόρηση πρέπει να περιέχεται στις εκθέσεις. Η διαφάνεια είναι βασικό στοιχείο. Να αυξηθεί η διαφάνεια. Θέλουμε λοιπόν ένα ρωμαλαίο MRV που να είναι καταλήτης για να ενθαρρύνει και να δώσει τη δυνατότητα και στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές να λαμβάνουν αποφάσεις που να αυξήσουν την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, η λειτουργική αποτελεσματικότητα στα μέσα μεταφοράς πολλές φορές ε, σχετίζεται με το λόγο μεταξύ κατανάλωσης ε, καυσίμων και της υπηρεσίας που παρέχεται, δηλαδή της μεταφοράς του φορτίου ε, ανάλογα με την κατανάλωση. Άρα δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε το φορτίο που μεταφέρεται. Δεν είχαν αποτελέσματα τα MRV. Η λειτουργική αποτελεσματικότητα και η σύγκριση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των πλοίων είναι φυσικά περίπλοκη. Χρειάζεται κάποια πείρα όμως αυτοί που ενεργοποιούνται στο ναυτιλιακό τομέα είναι συνηθισμένοι να συλλέγουν και να χορηγούν πληροφόρηση για να λαμβάνονται σωστά οι αποφάσεις. Τα στοιχεία για το φορτίο που, που, που προτείνονται στο MRV δεν νομίζουμε ότι είναι ευαίσθητα για τις επιχειρήσεις γιατί θέλουμε ετήσια συνολικά στοιχεία και δεν θέλουμε στοιχεία για ε, ε, μεμονωμένα ταξίδια. Δεν θα μπορούν λοιπόν όσοι έχουν πρόσβαση να πάρουν πληροφόρηση για συγκεκριμένα φορτία, διαδρομές, ε, ιδιοκτήτες φορτίων κτλ. Ήδη ε, απαιτούνται από ε, διάφορα νομικά συστήματα τα στοιχεία αυτά για λόγους ασφαλείας. Και το τμήμα επιτήρησης του ΕΜΑΒ σε μεγάλο βαθμό ήδη υπάρχει. Αν εξετάσουμε τώρα τι συζητήσεις γίνονται στον ΑΕΜΟ για την λειτουργική ενεργειακή αποτελεσματικότητα και προδιαγραφές στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν θέματα φορτίου. Να εξαιρέσουμε το φορτίο από το πεδίο εφαρμογή του MRV της Ένωσης θα καθιστούσε πολύ δύσκολο για την Ένωση να παίξει ηγετικό ρόλο σε αυτή τη συζήτηση. Θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα εμπόδιο για τη συμμετοχή μας στη διεθνή συζήτηση. δημοσίευση ανωνύμων στοιχείων για κάθε πλοίο. Την... Και εδώ η αύξηση της διαφάνειας είναι βασικό στοιχείο για ένα MRV που να μπορεί να λειτουργήσει μόνο του. Ναι, μπορεί να, ανεβάσει, να αποτελέσει βάση και για άλλα στοιχεία πολιτικής, αλλά το MRV από μόνο του θα πρέπει να μας επιτρέπει να δώσουμε τα αναγκαία κίνητρα στον κλάδο για να μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους μας μόνο αξιόπιστα και συγκριτικά στοιχεία για την ενεργειακή αποδοτικότητα θα διασφαλίσει να λαμβάνονται αποφάσεις ε, επιχειρηματικές όπως ναύλωση ή αγορά μεταχειρισμένων πλοίων αξιοποιώντας αυτά τα στοιχεία. Τα στοιχεία που έχουμε τώρα δεν είναι ούτε αξιόπιστα ούτε συγκρίσιμα. Δεν έχουμε προδιαγραφές στον τομέα αυτό σήμερα οι, τα, οι προδιαγραφές λειτουργικής αποτελεσματικότητας που συζητάτε στον IMO βασίζεται σε δύο αρχές. Να χρησιμοποιούμε ε, ελάχιστα επίπεδα για κατηγορίες πλοίων ή για συγκεκριμένα πλοία. Η δεύτερη αντίληψη θα σήμαινε να γίνεται υποβολή εκθέσεων και δημοσίευση στοιχείων αναπλοίο. Πολύ νωρίς είναι για να εξαιρέσουμε μία από τις δύο εναλλακτικέ και οποιαδήποτε πρόορη απόφαση ενωσιακό επίπεδο μπορεί να θέσει εν κινδύνο τις γενικότερες συζητήσεις και το σημαντικό ρόλο της Ένωσης σε αυτές τις συζητήσεις. Τώρα να διευρύνουμε το φάσμα και για άλλους ρηπαντές. Εμείς θέλαμε να είμαστε περιορισμένοι και ρεαλιστές. Θέλουμε να έχουμε μία εικόνα για την αυτιλία μας στην Ένωση. Θέλουμε να είναι αποτελεσματικό το σύστημά μας και να μην είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατικό. Διότι ακούμε για αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, ότι υπάρχουν πολλές πιέσεις λόγω και της οικονομικής κρίσης που παρατηρούμε και στην ε, ναυτιλία. Οι εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα αναπλοίου μπορούν να υπολογιστούν με βάση τις πληροφορίες για την κατανάλωση καυσίμων. Αυτά τα στοιχεία τα έχουμε σχεδόν ε, για όλα τα πλοία ήδη η απλούστερη μέθοδος παρακολούθησης που να βασίζεται με τα έγγραφα που έχουμε ήδη για την κατανάλωση καυσίμων δεν θα λειτουργήσει όμως για τα οξύδια του αζότου. Άρα αυτά τα στοιχεία δεν θα μας προσφέρουν ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία από τις αναλύσεις και μελέτες που έχουμε ήδη. Αν βάλουμε και άλλες ουσίες τώρα σε αυτό το MRV θα έπρεπε να βάλουμε ιδιαίτερα δαπανηρούς μετρητές αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται αυτοί οι μετρητές και έχουμε ήδη θετικές εμπειρίες από αυτούς, αλλά είναι κάπως πειραματική ε, η λειτουργία τους, για παράδειγμα, όταν ε, έχει φουρτούνα. Δεν έχουμε παρκή πληροφόρηση για το κόστος τους, λοιπόν. Έχουμε κάποιους υπολογισμού που μοιάζει να λένε ότι οι μετρητές για το άζωτο θα μπορεί να σήμαιναν πάνω από 100.000 ευρώ ανά σκάφος, ανά πλοίο. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι δυσχερές. Αλλά αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η παρακολούθηση όλων των ρηπαντών είναι πολύ σημαντική. Και γι' αυτό να το συζητήσουμε. Είμαστε ανοιχτοί για μια πιο πλήρη αντιμετώπιση εφόσον και όταν οι τεχνολογίες θα είναι διαθέσιμες σε λογικό κόστος. Και η Κομισιόν γενικά έχει ε, ανοιχτή στάση απέναντι σε αυτό. Τώρα, η δημιουργία ενός κατώτερου κατοφλίου που προτείνει ο εισηγητής και κάποιες γνωμοδοτήσεις. Το όριο των 5.000 τόνων είναι καλό σημείο διαχωρισμού κατά τη γνώμη μας. Και είναι ε, σωστή αναλογικότητα. Αν μειώσουμε αυτό το κατόφλιο, θα πρέπει να καλύψουμε πάρα πολλά πλοία. Από 55% του στόλου όπως είναι τώρα, σε πάνω από 90% του στόλου. Και θα μας πρόσθεται μόνο 10% των συνολικών εκπομπών. Πολιτικά είναι λογικό να θέσουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο. Υπάρχει μια πρόταση από τον εισηγητή, ένα χαμηλότερο κατόφλιο θα ήταν ε, πιο συντονισμένο με τη συζήτηση των IMO. Ε, το χαμηλότερο όμως κατόφλιο θα αυξήσει και το κόστος για τον τομέα. Τώρα υπολογίζουμε ότι είναι στα 80 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορούσε να πάει στα 148 εκατομμύρια. Θα είχε λοιπόν μεγαλύτερη επίπτωση στις μικρομεσαίες. Κάτι ακόμη. για τα σχόλια της κυρίας Μακάβαν και των Πρασίνων. Το 2008 το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κάλεσαν να υπάρξει πρόταση για μέτρα για να μειωθούν τα αέρια θερμοκηπίου από την αυθυλία ελήψη παγκόσμιας συμφωνίας και υπόθηκε ότι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο σύστημα εμπορίας εκπομπών για να προχωρήσουμε. Αλλά έκτοτε έχουν υπάρξει πολύ σημαντικέ εξελίξεις στον IMO μέσω της πρότασης MRV που συζητείται. Αυτή τη στιγμή οι εμπειρογνώμονες εργάζονται ιδιαίτερα έντονα. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο ένα τέτοιο σύστημα. Λόγω λοιπόν αυτών των συνδικών είναι σημαντικό η Ένωση να καταστεί σαφέ ότι είναι τμήμα αυτή τη ε, παγκόσμια συζήτησης ούτω ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε την ε, καλύτερη ε, εμπειρογνωμοσύνη και να συμμετάσχουμε με τον πιο επικοδομητικό τρόπο. Είναι σημαντικό λοιπόν να προτείνουμε ένα ρωμαλαίο και φιλόδοξο MRV. Έτσι μπορούμε και να συμβάλλουμε αλλά και να ηγηθούμε στις συζητήσεις των ΑΕΜΟ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αναλυτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις. Και τέλος, ο κύριος Κυλακάκης ως συζητητής. Παρακαλώ. Θα είμαι σύντομος για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, οι Αμερικανοί δεν περιλαμβάνουν το έργο μεταφορών ε, στο ε, τελευταία τους έγγραφα. Εάν φτιάξουμε το MRV με το έργο μεταφορών και μετά ο ΑΕΜΟ επιλέξει χωρίς, θα πρέπει είτε να αλλάξουμε το δικό μας MRV, βγάζοντας έξω το έργο μεταφοράς, το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο, είτε θα έχουμε δύο MRV, ένα παγκόσμιο και ένα ευρωπαϊκό, το οποίο θα ήταν λάθος. Ο άλλος τρόπος είναι πιο εύκολος. Εάν οι Αμερικανοί ή ο IMO αποφασίσουν όλοι ότι θα συμπεριληφθεί το έργο μεταφοράς, μπορούμε να τα αλλάξουμε. Διότι δεν θα είναι πολιτικά δύσκολο. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Δεύτερον, φυσικά, αν έχουμε όλα τα στοιχεία τα οποία θα παρέχονται επώνυμα, θα είναι αξιόπιστα, και συγκρίσιμα. Δεν αλλάζει τίποτα στη συγκρισιμότητα και στην αξιοπιστία των δεδομένων ε, εάν δεν έχουμε τα ονόματα. Αλλά το πλεονέκτημα είναι ότι δεν θα γίνονται επιθέσεις παραπλανητικές ε, σε μη αποδοτικές επιχειρήσεις ή πλοία όταν για πολύ καλούς λόγους, λόγω δρομολογίου για παράδειγμα ή λόγω καιρικών ε, δυσκολιών δεν μπορούν να είναι ενεργειακά αποδοτικά κάποια συγκεκριμένα πλοία. αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα, ευρετήριο, ένα δίκτυο ε, ενεργειακής απόδοσης θα το ονομάσουμε έτσι. Ας, μην, ας είμαστε ειλικρινείς. Ας έχουμε ένα κανονισμό για την ενεργειακή απόδοση των πλοίων. Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε ένα πράγμα και κάτω από αυτό κάτι άλλο. Κατά την άποψή μου η ενεργειακή απόδοση είναι το πραγματικό ζήτημα. Εγώ πιστεύω στην αρχή ορυπένων πληρώνει. Αυτή η αρχή πρέπει να εφαρμοστεί. Εάν βασίσουμε όσα θέλουμε να κάνουμε στην ενεργειακή απόδοση, πετάμε στα σκουπίδια την ε, αρχή του ορυπένων πληρώνει. Πιστεύω ότι αυτός ο κανονισμός προσπαθεί να θεωρήσει ότι η ενεργειακή απόδοση είναι το κύριο ζήτημα με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί κάποια στιγμή η αρχή ορύπανο πληρώνει και εγώ πιστεύω ότι αυτή θα ήταν λάθος οδός. Γι' αυτό το λόγο το υποστηρίζω τόσο στενάρα. Τέλος, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή. δεν είναι το 10% το θέμα. Το πρόβλημα είναι η στρέβλωση. Το γεγονό είναι ότι αν αποκλείσουμε όλα τα μικρότερα πλοία, τότε θα έχουμε ένα κόμβο, για παράδειγμα τη Μεσόγειο, όχι στο Βόρα, γιατί δεν υπάρχει κόμβος, αλλά στη Μεσόγειο θα υπάρχει ένας κόμβος και όσοι έχουν εξαιρεθεί θα, θα, θα εξαιρούνται Όλα τα πλοία, τα μικρά που εξαιρούνται από τους βόρειους κόμβους θα πηγαίνουν στο νότο, στα λιμάνια του νότου και εκεί θα μεταφέρουν φορτία. Δεν θέλουμε αυτό όμως. Δεν θέλουμε στρέβλωση τέτοιου είδους. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει το πεδίο εφαρμογής να είναι ευρύτερο. Ευχαριστώ. Έχω μια αίσθηση ότι έχω ξαναδεί την κατάσταση. Είναι η ίδια συζήτηση που είχαμε και νωρίτερα για τους κόμβους. Θα ξανακάνετε τη συζήτηση. Οπότε, κλείνουμε τη συζήτηση. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών 4 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Οι οποίες θα συζητηθούν στις 22 Ιανουαρίου ως Επιτροπή θα ψηφίσουμε στις 30 Ιανουαρίου και ελπίζουμε τον Απρίλιο όπως ελπίζουν και πολλοί άλλοι συγκητές να υπάρξει λύση και ψηφοφορία κατά την πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή, ευχαριστώ για όσους ε, εκπροσώπησαν τους ε, σκιώδεις. Θα τα πούμε με τον πρώην Υπουργό της Πολωνίας που τώρα είναι αρμόδιος μόνο για το κλίμα και είναι ε, εκπρόσωπος ε, των διαπραγματεύσεων ΚΟΠ από τις 3 ε, ώρα και μετά. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Μέχρι τότε χαίρετε.